Yeah. No. Okay. Yeah. Yeah. Good afternoon, dear colleagues. Καλησπέρα σας συνάδελφοι. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. And if there are no changes proposed. Αν δεν υπάρχουν αλλαγέ για την ημερήσια διάταξη, εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Δεύτερο σημείο στην ημερήσια διάταξη, ανακοινώσεις της Προέδρου. Σημείο 2.1. Ανακοινώσεις για τις συστάσεις των συντονιστών της συνεδρίας της 11 Απριλίου και Εκεί οι συντονιστές αποφάσισαν να υποβάλουν τροπολογίες στην έκθεση επιτροπή Επιτροπής Απασχόλησης για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Αναπηρίας και να το δώσουμε στο ΕΛΚ. Επίσης, να υποβάλουν τροπολογίες στην έκθεση ΠΕΤΗ για την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια του 2017 και να ανατεθεί στην ομάδα της ΓΟΕ. Να διατυπώσει μια προφορική ερώτηση με ψήφισμα για τους ε, γάμους ανηλίκων και να την εγκρίνει στην Επιτροπή ΦΑΜ στη διάρκεια του Μαΐου και να καλέσουμε την κυρία Μανουέλα Σβέσικ, ε, Γερμανίδα Υπουργό Οικογενειακών Υποθέσεων Ηλικιωμένων Γυναικών και Νεολαίας, ε, σε μια μελλοντική συνεδρία της Επιτροπής μας. Στη συνεδρίαση της 25ης Απριλίου οι συντονιστές αποφάσισαν να υποβάλλουν τροπολογίε για να διατυπώσουν τη θέση της για την καταπολέμηση των ανισοτήτων ω μοχλό για την όθηση της δημιουργία θέσεων εργασία και τη ανάπτυξη και να ανατεθεί στην ομάδα του ΕΛΚ. Να γίνει αποστολή στο Μαρόκο από 18-20 Σεπτεμβρίου του 2017 και επικεφαλής αποστολής θα είναι η κυρία Λεγκρίπ. Να καλέσουμε εκπρόσωπο του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών σε μία από τις μελλοντικές συνεδριάσεις Επιτροπής μας. Σημείο 2.2 για ε, τις υπόλοιπες ανακοινώσεις, η Επιτροπή ΔΕΒΕ αποφάσισε να οργανώσει μια συζήτηση για τον κανόνα της ολικής ε, φήμωσης, τον Global Gag Rule. Η συζήτηση αυτή θα γίνει στη συνεδρία της Επιτροπής ΔΕΒΑ ε, στις 29 Μαΐου, ημέρα Δευτέρα, και οι συντονιστές αποφάσισαν να καλέσουν την Επιτροπή Γυναικών, Προϋπολογισμών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θα λάβετε όλη η πρόσκληση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τη συμμετοχή σας. Αυτές λοιπόν ήταν οι ανακοινώσεις του Πρόεδρου και τώρα περνάμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης στην ηλεκτρονική ψηφοφορία. Συνάδελφοι, είστε έτοιμοι για την ψηφοφορία? Έχετε τις κάρτες σας. Ωραία.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 κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Σημείο 4 τώρα. Σχέδιο έκθεσης ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για να ε, προλάβουμε το κενό στις συντάξεις μεταξύ των φίλων. Η συγκήτρια Κωνσταντς Λεγκρίπ από το ΕΛΚ. Συμβαστική τροπολογία 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να κάνουμε μια επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε λοιπόν την τροπολογία 106. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμών 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 110 υπέρ. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να κάνουμε επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Vote is closed. Πέραση της Απορρίπτεται. 174 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. 174 δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία για την 174 δεύτερο τμήμα πέρασε ψηφοφορίας. Μισό λεπτό. Your card function. Δεν δούλεψε η κάρτα σας. Όχι, δεν δούλεψε. Υπέρ ή κατά ψηφίσατε. Πώς ψηφίσατε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Είμαστε κατά. Ψηφίζει.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 Compromise 3 in Χωρί μικρόφωνο, πρόεδρο. Συμβαστική τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. 128 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 134 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 4 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Διακόσια υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Για τη 240 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρες τη ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ζητώ συγγνώμη. 143 υπέρ, σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία, της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 145 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία. 145. Ψηφίζουμε την 145. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 148. Υπέρ. Κατά. Συνάδελφοι, πρέπει πάλι να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 147 υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία για την 147. Πέρασε της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Έμπλ 33 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά αποχές πρέπει να επαληθεύσουμε ζητώ συγγνώμη άρχεται η ψηφοφορία πέρασε της ψηφοφορίας απορρίπτεται έμπλε 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Επαλήθευση, εντάξει, να επαληθεύσουμε. Έμπλη 34, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρασε ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Με μία ψήφο διαφορά. All electronic. No, we will look. No, no. Sometimes, yeah, yeah, yeah, yeah. Okay. Amendment 100. Τροπολογία 150 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Επαλήθευση για την 150. Επαλήθευση για την 150. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε η ψηφοφορία. Adopted. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 146 υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση τη ψηφοφορίας, εγκρίνεται. 167 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ. Κατά αποχές πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε της ψηφοφορία. Απορρίπτεται. 179 υπέρ. 179 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι γκρίνεται, αλλά πρέπει να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 180 υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαλήθευση παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 234 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 185 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 187 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 200, υπέρ, κατά, αποχές, επαλήθευση παρακαλώ, άρχεται την ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμ... Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ. Θέλετε να επαληθεύσουμε τη 13? Ε, εντάξει, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 2.19 υπέρ, κατά, αποχές, επαλήτευση. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 220 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 222 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 224 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 223 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Έμπλη 17, υπέρ. Σελίδα 18 στο δικό μου τον κατάλογο, έμπλη 17 υπέρ. Κατά, αποχές, πρέπει να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Έμπλη 28 υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Επαλήθευση. Άρχεται ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Έμπλικος 29 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογική έκθεση 1 της έμπλη υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 2 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ έκθεση 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Να το επαληθεύσουμε, ναι, άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed is rejected. Πέραση της ψηφοφορίες απορρίπτεται. Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Έμπλ, αιτιολογική έκθεση 6, 3 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 4 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Έμπλ 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να το επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία, πέραση της ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Έμπλ 10 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έμπλετ 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 9 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να το επαληθεύσουμε, άρχεται η ψηφοφορία, πέρασε η ψηφοφορία. It's adopted. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17 υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας την ελέγξουμε ηλεκτρονικά λοιπόν. Τροπολογία 16. Πέραση της Επαναλαμβάνουμε λέει ο Πρόεδρος. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν για την τροπολογία 16 την ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 18 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εμπλ Εν. τμήματική ψηφοφορία σε τρία τμήματα. Επί του πρώτου ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μήμα δεύτερο ψήφι περ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τρίτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές Ας ελέγξουμε λοιπόν. Άρχεται η ψηφοφορία για το τρίτο τμήμα. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Συμβαστική τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. εγκρίνεται. Τροπολογία 38 ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 37 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 39 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έμπλ C υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται νομίζω αλλά την ελέγξουμε την Έμπλ Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Έμπλυντή D ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Έμπλ B, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 22. Α, όχι, να ελέγξουμε. Να ελέγξουμε την Έμπλ B, άρχιτη ψηφοφορία. Πέρας, εγκρίνεται. Με διαφορά μια ψήφου. Είναι δύσκολο. Συμβασική τροπολογία 22. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω πως απορρίπτεται αλλά στην ελέγξουμε. Τροπολογία 42. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 52 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 62-63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται. 65 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτονται. 67. Να ελέγξουμε την τροπολογία 65. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 66 περ κατά αποχές απορρίπτεται. MPG σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 28 ψήφι υπέρ Θέλετε να ελέγξετε τη συμβαστική 27, οπότε την ελέγχουμε. Άρχη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28 ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την ελέγξουμε. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για τη συμβαστική τοπολογία 29. Πέραση της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 86 λοιπόν ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέραση της ψηφοφορίας απορρίπτεται 87 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε την 87 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 88 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές ας ελέγξουμε την 96 ηλεκτρονικά πέρασε της φοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. Ελέγχουμε λοιπόν ηλεκτρονικά. Πέραση της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε επί του συνόλου της πρότασης ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. Άρχεται η ψηφοφορία. The is closed. Πέραση της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε άλλες φοροφορίες. Ε, θα θέλαμε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 Uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση σημείο 5 στην ημερήσια διάταξη 10 βασικά μηνύματα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα τα βρείτε στα έγγραφα της συνεδρίασης, τα δέκα βασικά μηνύματα αυτά, τα σχέδιά τους, όπως προτάθηκαν από τις πολιτικές ομάδες. Υπάρχουν τρεις κύριες προτεραιότητες. Στρατηγική για την ισότητα των φύλων, συνδυασμό επαγγελματική και δυτικής ζωής και βία με βασί το φύλο και επτά ακόμη σημεία γυναίκε σε διοικητικά συμβούλια και σε διαδικασίε λήψη αποφάσεων, το συνταξιοδοτικό χάσμα λογοφύλου, εμπορία ανθρώπων, ισότιμη μεταχείριση στην απασχόληση και στην εκπαίδευση, το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος λογοφύλου, η συνεκτήμηση της διάστασης του φύλου στις ευρωπαϊκές πολιτικές και σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και δικαιώματα. Τα δέκα βασικά μηνύματα αυτά θα εγκριθούν στις 11 Μαΐου στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Οπότε αν δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο σχετικά με τις προτάσεις των πολιτικών ομάδων θα ψηφίσουμε την επόμενη φορά και τώρα έχουμε εδώ μαζί μας την Επίτροπο Γιώργοβα στις 4 η ώρα, οπότε έχουμε κάποιο καιρό για διάλειμμα, αλλά παρακαλώ ας είστε εδώ στις 4. Otherwise, Υπότιτλοι AUTHORWAVE

στο κατήχη παλάτι. Okay, okay.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

Συνεχίζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, την ε, συνεδρίασή μας με το επόμενο σημείο της μέρης σας διάταξης ε, με την Επίτροπο κυρία ε, Γιούροβα, Επίτροπο για ζητήματα δικαιοσύνης και ισότητας των φίλων. Σας ευχαριστούμε κυρία κύριε που βρίσκεται σήμερα εδώ στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πάντοτε καλωσορίζουμε τη συμμετοχή σας στις εργασίες μας, ειδικότερα καθώς δεν είχαμε τη δυνατότητα να το πράξουμε και αρκετό δηλαδή να σας συναντήσουμε εδώ ε, στην Επιτροπή ΦΑΜ. Ο διαρθωμένος διάλογος είναι πολύ σημαντικός για μας, όπως γνωρίζετε, οπότε σας ευχαριστώ πολύ ε, για την προσέλευση σήμερα εδώ και σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστούμε κυρία Πρόεδρε, ευχαριστούμε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Βρισκόμαι με την μου σήμερα εδώ και πραγματικά ε, το εννοώ ειλικρινά. Είναι τιμή μου να βρίσκομαι σήμερα εδώ γιατί αποτελεί μια πολύ καλή ευκαιρία όχι μόνο να πληρώσω τα καθήκοντά μου απέναντί σας ως προς ε, δηλαδή την ευθύνη ε, ως επίτροπος απέναντι στο Κοινοβούλιο αλλά και προκειμένου να ακούσω τις δικές σας ιδέες, τα ενάβασματα για σκέψη σας καθώς μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι κάνουμε κύκλους προσπερνούμε δηλαδή ο ένας τον άλλο σε ό,τι αφορά τις σκέψει μας. Οπότε όποτε σας βρίσκω, μέρο και στι ε, διάφορες ε, ε, επιτροπές και στην Ολομέλεια, πάντοτε προσπαθώ να προβαίνουμε σε ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά τα ζητήματα ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Νομίζω πως σήμερα είναι μια ιδιαίτερα καλή χρονική συγκυρία για μια τέτοια συζήτηση, γιατί πριν από λίγο έγινε η παρουσίαση του πακέτου σε ό,τι αφορά την ισορροπία μεταξύ εργασιακή και ιδιωτική ζωή σε σχέση πάντοτε και με την σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη. Οπότε νομίζω πω έχουμε πολλά να συζητήσουμε σήμερα. Θα κάνω μια σχετικά σύντομη παρουσίαση από τη δική μου πλευρά για να προχωρήσουμε στη συνέχεια στη συζήτηση. Λάβαμε λοιπόν νεότερα δεδομένα ε, στο πλαίσιο τη έκθεση για την ισότητα μεταξύ των δύο φύλων που δημοσιεύθηκε το Μάρτιο και τα ε, βασικά νούμερα εδώ είναι τα εξή. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στην ε, αγορά εργασίας, δηλαδή αποτελούν το 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού, αλλά μόνο το 65% των γυναικών συμμετέχουν στην εργασιακή αγορά, ενώ το 75% των ε, αντρών συμμετέχουν στην εργασιακή στην αγορά εργασίας και συχνά βέβαια έχουν το πρόβλημα της φροντίδας ε, των παιδιών και ένας ακόμα σημαντικός ε, παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες είναι πολύ πιο εκτεθειμένε ε, στην ένδια από ότι οι άνδρες. Και εδώ έχουμε να κάνουμε με μια αστοχία αν θέλετε της αγοράς η οποία μας κοστίζει το 2,8% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετησίως. Αυτή δηλαδή η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας μας κοστίζει λοιπόν ετησίως 2,8% του ΑΕΠ μας γύρω στα 370 δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν αυτό ε, ο αριθμός. Ενώ και πραγματικά ε, δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό το νούμερο όταν ε, το διάβασα για πρώτη φορά και απευθύνθηκα στους υπεύθυνους από την πλευρά της που συνέταξαν δηλαδή την έκθεση και μου εξήγησαν ποια μεθοδολογία εφάρμοσαν και πώς προέκυψε δηλαδή αυτό το νούμερο και πράγματι έτσι ήμουν σε θέση να ελέγξω ότι πρόκειται και για μια πολύ συντηρητική εκτίμηση. Ε, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή και το σχετικό πακέτο που προτείναμε, νομίζω πω ε, χρειάζεται να συζητήσουμε για την ανισότητα ταυτόχρονα και για τι ίσε ευκαιρίε, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει να μιλήσουμε και για του οικονομικού παράγοντε ε, και την αστοχία, αν θέλετε, εδώ, σε αυτό το επίπεδο τη αγορά εργασία τη Ευρωπαϊκή Ένωση και το τι σημαίνει αυτό ε, ως απώλειες οικονομικές. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ένδια και την υποπροσώπηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, αυτό που θα πρέπει να λάβουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας είναι το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούν σήμερα ε, το 60% των αποφύτων των πανεπιστημίων και κατά συνέπεια ε, τα ταλέντα τους, τα προσόντα τους θα πρέπει να αξιοποιηθούν καλύτερα από την κοινωνία τους ταυτόχρονα. Υπάρχουν και περισσότεροι πατέρες που θέλουν να ε, περνούν περισσότερο χρόνο ε, με ε, τα παιδιά τους. Και επίσης η γενιά των millennials όπως λέγεται θέλουν περισσότεροι να λαμβάνουν υπόψη τους τον παράγοντα της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτικής ζωής όταν επιλέγουν τον εργοδότη της. Από εκεί και μετά έχουμε το φαινόμενο της γύρανσης του πληθυσμού που σημαίνει ότι όλο και περισσότερες οικογένειες θα χρειάζεται να φροντίσουν τους συλλογιωμένους συγγενείς τους και ταυτόχρονα η ψηφιακή επανάσταση καθιστά δυνατές και καθιστά πραγματικότητα τις ε, ψηφιακές, τους ψηφιακούς όρους εργασίας σε μια σειρά από Άρα λοιπόν όλες αυτές οι διαστάσεις ήταν εκείνες οι οποίες λάβαμε υπόψη μας στο πλαίσιο της προπαρασκευής ε, των νομοθετικών και μη νομοθετικών ε, προτάσεων και εργαλείων που προτείνουμε για την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής γνωρίζουμε ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε λύσεις σε ό,τι αφορά το σύγχρονο τρόπο ζωής ε, και να τη συνδυάσουμε με καλύτερη παροχή υπηρεσιών, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα δεύτερα μέλη, αν θέλετε, δηλαδή πέρα από τον ε, κύριο, ε, το κύριο άτομο του νοικιού κορκυριού που φέρνει το εισόδημα, να λάβουμε υπόψη μας και τα άλλα μέλη της οικογένειας που μπορούν να προσφέρουν εισόδημα. Το πακέτο λοιπόν αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς σήμερα αποτελείται από νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα. Δεν δηλαδή κάνουμε προτάσεις, προτάσεις νομοθετικέ. Όχι, πρόκειται για ένα σύνολο, μια δέσμη προτάσεων, συνεκτικό ελπίζω. Η ε, πρόταση λοιπόν ε, εξυγχρονίζει το πλαίσιό μας, ώστε να ανταποκριθούμε στα προβλήματα που έχουμε, δηλαδή έλλειψη αποσμίωσης, έλλειψη ευελιξίας και μη ε, δυνατότητα μεταφοράς των διαφόρων προσόντων και προσπαθούμε να διασφαλίσουμε και να εξυγχρονίσουμε τα διάφορα εγγυημένα δικαιώματα τόσο για άντρε ε, και γυναίκε. Και σεβόμαστε πλήρω τι ατομικέ ελευθερίε ε, των γυναικών, των οικογενειών και δεν ε, ε, σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί εμπόδια στα κράτη-μέλη στην υιοθέτηση ακόμα αυστηρότερων κριτηρίων. Και εδώ θα πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Αυτό που κάνουμε δηλαδή εμεί εδώ με αυτή την πρόταση είναι να θέτουμε ελάχιστα κριτηρία. Σε ό,τι αφορά τώρα την ευελιξία τη γονική άδεια, θέλουμε μια, ε, ε, έναν εξυγχρονισμό των σχετικών διατάξεων σε ό,τι αφορά την μερική άδεια και σε ό,τι αφορά την δυνατότητα για την ε, λήψη της γονικής άδεια προτείνουμε την αύξηση από 8 σε 12 έτη και επίσης ε, σε ό,τι αφορά την, ε, την, την αποζημίωση για την γονική άδεια προτείνουμε αυτό το non-transferability, την αρχή του non-transferability, τέσσερις μήνες δηλαδή για τον δεύτερο γονέα και και ε, άδεια ασθενεία και για του δύο γονεί. Επίση, ε, προτείνουμε έναν εξεχρονισμό σε ό,τι αφορά τη γονική άδεια για του πατέρε για τα νεονά, δηλαδή 10 ημέρε μεταποδοχών. Από εκεί και μετά. Για να διευκολύνουμε ε, την καλύτερη, ε, το καλύτερο διαμερισμό μεταξύ των μελών της οικογένειας. Ε, προτείνουμε πέντε ημέρες άδεια μεταποδοχών, ώστε να επιστρέψουμε, επιτρέψουμε και στους άντρες και στις γυναίκες να προσαρμόσουν το εργασιακό τους πρόγραμμα και αξιοποιούμε και το δικαίωμά τους να αξιώσουν ευέλικτες ευέλικτο προγραμματισμό του ωραρίου εργασία τους ε, και για τα συγκεκριμένα τους εξαρτώμενα πρόσωπα και ε, σε αυτό το πλαίσιο προτείνουμε και μη νομοθετικές ε, δράσεις. Αλλά προτού περάσω σε αυτές τις μη νομοθετικές προτάσεις θα ήθελα να σας δώσω κάποιες περισσότερες λεπτομέρειες σε ό,τι αφορά αυτές τις μη νομοθετικές προτάσεις που κάνουμε. Νομίζω πως θα θυμόσαστε ε, την στιγμή όπου είχαμε αποσύρει από την πλευρά της Επιτροπής ε, την οδηγία για την μητρική άδεια γιατί είχε μπλοκαριστεί στο επίπεδο του Συμβουλίου και βέβαια ήδη η πλειοψηφία των κρατών μελών προέβλεπαν στην ομοθεσία τους τέτοιου είδους ε, μέτρα τα οποία δηλαδή περιλαμβάνονταν σε αυτήν την οδηγία για την πατρική γονική άδεια. Οπότε τώρα κάνουμε μια πρόταση με νομοθετικές με νομοθετικά στοιχεία, δηλαδή διάφορες νομοθετικές προτάσεις που θα αφορούν τις σχετικές άδειε όχι μόνο για τα νεονά, αλλά και ε, κάποιες διατάξεις σε ό,τι αφορά το δεύτερο γονέα, δηλαδή συνήθως ε, τον ε, πατέρα, για την ε, ψηλότερη εμπλοκή αυτού του δεύτερου γονέα στην ιδιωτική ζωή, στην οικογενειακή ζωή, προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας ε, τις ιδιαίτερες απαιτήσει, ε, όπως για παράδειγμα ε, γυναικών οι οποίες πρέπει να φροντίζουν ταυτόχρονα και τέκνα αλλά και ε, για παράδειγμα εξαρτώμενους γονείς τους ως της οικογένειας. Οπότε θεωρώ πως η συζήτηση που θα κάνουμε θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα και ε, όπως σας είπα, όλες αυτές οι προτάσεις συνοδεύονται και από μη νομοθετικού χαρακτήρα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνονται στο ίδιο πακέτο. Σε αυτές τις δράσεις λοιπόν αναφερόμαστε στη χρηματοδότηση και την παρακολούθηση ε, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εξαμήνου αυτών των δράσεων, ειδικότερα και συλλογή σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεδομένων, όπω και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και συνεχή παροχή καθοδήγηση στα κράτη-μέλη. Εκείνο που μπορώ να σα πω είναι ότι το εν πακέτο, ειδικότερα η μη νομοθετική πτυχή του αφορά ειδικότερα συνεργασία και ένταξη στις ε, βασικές ε, πολιτικές της διάστασης του φύλου ε, με τις διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί είχαμε τον Επιτροπό Πρόφστη, τον Πρόεδρο Τίμερμαντς, τον Κατάνεν και την Κούρινα Κρέτσου βέβαια η οποία είναι η θεματοφύλακας αν θέλετε των Ευρωπαϊκών Ταμείων και ο Γέρεμος συνέβαλε επίσης από την πλευρά του μέσω συστάσεων σε ό,τι αφορά την τροποποίηση των φορολογικών συστημάτων ε, στα κράτη-μέλη έτσι ώστε να ευνοούν ακριβώς ε, τις ε, οικογένειες. Τώρα, να περάσω σε κάποια παραδείγματα ως προς τις μη νομοθετικές αυτές δράσεις που σας ανέφερα. Θέλουμε να ενισχύσουμε την εφαρμογή της υφιστάμενης νομικής προστασίας σε ό,τι αφορά τις απολύσεις εγγύων γυναικών ε, και μητέρων ε, μέσω ειδικότερα εκστατιών ενημερωτικών για την ευαισθητοποίηση του κοινού. Επίσης, άλλο στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε ε, τους νέους μάλλον να ενθαρρύνουμε τη χρηματοδότηση των σχετικών υποδομών μέσω του Ταμείου για τις μακροπρόθεσμες τις υπηρεσίες μακροπρόθεσμης φροντίδας. Τώρα, σε ό,τι αφορά, επανέρχομαι στο ζήτημα, την προστασία των εγγύων ε, γυναικών και μητέρων, ε, μου είχατε Κάποιοι από εσά αναφέρει ότι θα θέλατε να υπάρξει μια ξεχωριστή νομοθετική πρόταση. Ωστόσο, η εν λόγω εγγύηση, η εν λόγω προστασία ήδη περιλαμβάνεται στη νομοθεσία. Εκείνο δηλαδή που διαπιστώσαμε είναι ότι απλώ δεν εφαρμόζεται η εν λόγω διάταξη. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, ένα από τα μέτρα που προτείνουμε είναι να ξεκινήσει ένα διάλογο με τις διευθύνσεις επιθεώρησης εργασίας και τις διάφορες ε, επιβολής εδώ της εργασιακής νομοθεσίας στα κράτη-μέλη, οι οποίες είναι αρμόδιες για την ε, εποπτεία της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε να τους ασκήσουμε πιέσεις προκειμένου ακριβώς να εφαρμόζεται αυτή η διάταξη σε ό,τι αφορά την προστασία των εγγύων ε, μετρών από απολύσει. Τώρα, σα αναφέρθηκα και στη χρηματοδότηση από το Ταμείο μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, αλλά υπάρχουν και τα κλασικά εντό εισαγωγικών ευρωπαϊκά ταμεία τα μπορούν, να, ε, μπορούν να αξιοποιηθούν για την παροχή πιο προσιτών τιμολογιακά υπηρεσιών ε, σε πατέρες και φροντιστές για παράδειγμα μέσω γρεφονιπιακών σταθμών ή μέσω καταστάσεων στέγασης ε, για ηλικιωμένους ε, που ε, έχουν ως στόχο ακριβώς να, να δώσουν περισσότερες δυνατότητες να διευκολύνουν την παροχή φροντιδα σε τόσες οικογένειες. Άρα λοιπόν αυτή η αξιοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων για τέτοιου είδους δαπάνες αποτελεί μια καινοτομία γιατί οι κοινωνικές υπηρεσίες ανέκαθεν αποτελούσαν ή γίνονταν κατανοητές στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ένας τομέας δημοσίων επενδύσεων. Όμως εμείς θέλουμε να δώσουμε ε, περισσότερες δυνατότητες για έργα εδώ τύπου PPP, δηλαδή εταιρικών σχέσεων ιδιωτικού δημοσίου τομέα, αλλά και δυνατότητες ε, κοινωνικού επιχειρήν, social entrepreneuring, ε, σε ό,τι αφορά ειδικότερε οντότητε και επιχειρήσει και μη κυβερνητικέ οργανώσει, γιατί και αυτές ακριβώ οι φορεί μπορούν να συμμετάσχουν στη δημιουργία αυτών των σε ποιότητας υπηρεσιών για τι εν λόγω οικογένειε. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τι δυνατότητε χρηματοδότηση των μη νομοθετικών δράσεων. Καθώς ε, αναμένατε για αρκετό καιρό αυτό το πακέτο με υπομονή μάλιστα, το γνωρίζω αυτά που πλευρά του Κοινοβουλίου, αναμένω μεγάλο ενδιαφέρον τη σημερινή συζήτηση που θα γίνει γιατί να βέβαια ότι υπάρχουν πολλές καλές ιδέες και σχόλια τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στην περαιτέρω εργασία που θα κάνουμε σε σχέση με αυτό το πακέτο. Η νομοθετική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει. Τα μη νομοθετικά μέτρα από εκεί και μετά ε, είναι δυνατόν να ξεκινήσουν άμεσα και έχουμε μία σειρά από περιθώρια εδώ ευελιξία σε ό,τι αφορά την εφαρμογή, τον τρόπο εφαρμογή αυτών των μη νομοθετικών μέτρων. Ένα από του στόχου αυτού του πακέτου τη οροπία μεταξύ επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου είναι ακριβώ η αντιμετώπιση του τη μισθολογική ανισότητα μεταξύ των φύλων και η καταπολέμηση τη ένδυα στι γυναίκε με βάση δηλαδή και συνέχεια την ε, σύσταση σε ό,τι αφορά την ενίσχυση των αρχών για την ισότιμη, τις ε, ισότιμες αμοιβέ και την διαφάνεια σε ό,τι αφορά αυτές τις αμοιβέ, θα προβούμε και στην ε, πρόταση ε, περαιτέρω μέτρων σε αυτούς τους τομείς. Οπότε θα σας αναφέρω πώς θέλουμε να συνεχίσουμε για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος. Διότι πρόκειται για ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα αρκετές πηγές οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές αλλά με διαφορετικό τρόπο και αρκετά ισχυρές. Πρέπει να τα συζητήσουμε λοιπόν περαιτέρω, μπορούμε και να τα συζητήσουμε εδώ στη διάρκεια να σας πω και δύο λόγια για το πώς ε, θα προχωρήσουμε για την καταπολέμηση της βίας ε, εναντίον των γυναικών με καλύτερη οικονομική ανεξαρτησία για τις γυναίκες. Ο στόχος μας είναι να συνεισφέρουμε και στη μείωση των ανησυχητικών στοιχείων που έχουμε για τη βία, την έμφυλη βία. Και φυσικά γνωρίζετε ότι τα στοιχεία σοκάρουν, διότι Έχουμε την πιο πρόσφατη έρευνα η οποία καταδεικνύει ότι η στάση ε, έναντι του προβλήματος είναι εντυπωσιακή. Ε, περίπου το 25% ένας στους τέσσερις λοιπόν από αυτούς που απάντησαν ε, είπαν ότι συχνά οι γυναίκες είτε επινοούν είτε υπερβάλλουν στις καταγγελίες τους και ένα 17% υποστηρίζει ότι η βία κατά των γυναικών ορισμένες φορές προκαλείται από το θύμα. Ε, αυτό έρχεται να συμπληρώσει τα στοιχεία τα οποία είχαμε ήδη πριν από ένα χρόνο για τον τρόπο με τον οποίο ε, εμφανίζεται το φαινόμενο, πόσο συχνό είναι και πόσα θύματα έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών εξακολουθεί να είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό από τις κοινωνίες μας και θεωρείται φυσιολογικό ή και αναπόφευκτο. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένας από τους παράγοντες που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και να έχουμε κατά νου ε, σε ό,τι κάνουμε για τον τομέα αυτό. Με τις έρευνες αυτές ε, ταυτόχρονα ξεκινήσαμε και ε, μία σειρά από δράσεις για να εξαλείψουμε τη βία κατά των γυναικών το 2017. Προς το παρόν προσπαθούμε να συνδέσουμε και να υποστηρίξουμε τους ενδιαφερομένους προκειμένου να υπάρξει και ε, ανταλλαγή καλών πρακτικών ε, μεταξύ τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δόθηκαν 12 επιδοτήσεις σε εθνικές αρχές για να συγχρηματοδοτήσουν προγράμματα για την ανάπτυξη και εφαρμογή πρακτικών και στοχευμένων πληροφοριών, εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που στόχο έχουν να καταπολεμήσουν τη βία κατά των γυναικών και ε, εκστρατείες ευαισθητοποίησης. Ε, επίσης, ολοκληρώνεται τώρα η διαδικασία επιλογής ε, για τη χρηματοδότηση οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Ήμουν ιδιαίτερα ικανοποιημένη διότι η Μαλτέζικη Προεδρία έκανε μια διάσκεψη για τη βία κατά των γυναικών μέσα στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και είχαμε και τη δυνατότητα να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλον. Αναφερθήκαμε στο θέμα της βίας των γυναικών, προσπαθούμε να το ε, συμπεριλάβουμε σε άλλες οριζόντιες πολιτικές. Συνεργαζόμαστε με αρμόδιες οργανώσεις ε, και με τον επιχειρηματικό τομέα ακόμα για να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε τους πάντες. Διότι όπως σας είπα αυτό είναι πρόβλημα της κοινωνίας και επομένως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από διάφορους διάβλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εκτός, ε, μία στη Γεωργία προσφάτως, για να μπορέσουμε να ε, επιστήσουμε την προσοχή των ενδιαφερομένων επί του ζητήματος και ε, ε, στη συνέχεια της χρονιάς θα διοργανώσουμε και ε, σεμινάρια αμοιβαία μάθησης για να εδραιώσουμε τις πολιτικές μας και θα υπάρξει και μια εκδήλωση εδώ στο Κοινοβούλιο το Νοέμβριο, την οποία περιμένω με ανυπομονησία. Ε, το ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο ε, συμπεριλαμβανομένης και της οδηγίας για τα δικαιώματα των θυμάτων και το ευρωπαϊκό ένταλμα προστασίας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ε, η Eurostat έχει ξεκινήσει τις εργασίες της για να διεξάγει μια νέα έρευνα για τη βία για την έμφυλη βία, η οποία θα γίνει από τις Εθνικές Στατιστικές Υπηρεσίες με συντονισμό και στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος, κάτι αρκετά σημαντικό, να σας αναφέρω τις πρόσφατες εξαιρέσεις για την ε, προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, διάσκεψη της Κωνσταντινούπολης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έκανε προσπάθειες για επικοδομητικές συζητήσεις με το Συμβούλιο για να ξεκινήσει πολιτική συμφωνία για το θέμα αυτό και εσείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήσασταν ένας πάρα πολύ σημαντικός σύμμαχος της Επιτροπής αυτό με την συνεχή στήριξή σας ε, βρισκόμαστε πλέον στο τελικό στάδιο, το συμβιβαστικό κείμενο της ε, απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή της ε, διάσκεψης ε, του, της σύμβασης συγγνώμη, της Κωνσταντινούπολης πέρασε από την Κορεπέρ την προηγούμενη εβδομάδα. Η Επιτροπή θα διαβιβάσει το σχέδιο απόφασης στο Συμβούλιο για έγκριση τις επόμενες εβδομάδες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη συνεχή δέσμευσή σας για την καταπολέμηση της βίας ε, εναντίον των γυναικών, ιδιαίτερα της εισηγήτριες, την Άννα Κοράτσα Μπίλτ και την Σιλβί Μπονεφουά, Λοιπόν, για την ε, έκθεση για την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και για τη διοργάνωση σειράς ακροάσεων. Και για να ολοκληρώσω, να επιστρέψω ε, με τις γυναίκες τα διοικητικά συμβούλια. Πρόκειται για ένα θέμα που, πώς να σας το πω, ε, έχει ε, σταματήσει στο Συμβούλιο. Υπάρχει μια μικρή αργή πρόοδος σε εκπροσώπηση γυναικών στα διοικητικά συμβούλια ε, τα τελευταία πέντε χρόνια, αλλά γνωρίζουμε όλοι ότι παρόλο που έχει υπάρξει αυτή η πρόοδος, εάν υπάρξει νομοθεσία θα προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Υπάρχει ακόμα ένα στέλσο μειοψηφία στο Συμβούλιο, η οποία ελπίζουμε ότι θα αλλάξει μετά από τις γερμανικές εκλογές και θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε προκειμένου να πείσουμε τη νέα γερμανική αντιπροσωπεία και κάποια άλλα κράτη-μέλη να επανέλθουν στο θέμα αυτό. Σας ευχαριστώ για τη θερμή αντίδραση. Θα μπορούσα να σας λέω ιστορίες ολόκληρες για το τι ακριβώς κάναμε προκειμένου να πείσουμε τους Γερμανούς συναδέλφους και αντιλαμβάνομαι βεβαίως ότι ε, χρειάστηκε να δώσουν πάρα πολύ μεγάλη μάχη προκειμένου να εγκριθεί η εθνική νομοθεσία. Και εκεί ε, βρεθήκαμε εμείς με την οδηγία και το έτοιμα να συμμετέχουν και αυτοί ε, στην ομάδα των χωρών για την οδηγία για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια και κατάλαβα ότι δεν ήταν καθόλου ενθουσιασμένοι, δεν θα έπρεπε να ξανανοίξει η συζήτηση για την νομοθεσία. Χρειάστηκε λοιπόν να υπάρξει αμοιβαία συμφωνία για το πώς μπορούμε να το κάνουμε ώστε να μείνει ανέγγιχτος ο νόμος τους και να εγκρίνουμε και εμείς την οδηγία μας. Φυσικά ε, η διαδικασία αυτή κατέληξε σε αποτυχία. Πρέπει να περιμένουμε λοιπόν και να ξαναδοκιμάσουμε στη συνέχεια. Εν τω μεταξύ ανοίξαμε ένα δεύτερο μέτωπο και συζητάμε απευθεία με τις επιχειρήσεις και ε, με τη χάρτα της ποικιλομορφία, ε, το Business Europe και πολλές άλλες ε, οργανώσεις προκειμένου να μπορέσουμε να επιβάλλουμε κάποιες αρχές στα διοικητικά συμβούλια, στις επιχειρήσεις ώστε να έχουν περισσότερες γυναίκες σε κομβικές θέσεις. Και φυσικά δεν αναφερόμαστε μόνο σε υποπτικά συμβούλια αλλά και σε διοικητικά συμβούλια για να μπορούν να βρίσκονται και γυναίκες σε θέσεις εκτελεστικών διευθυντών ή ανωτέρων στελεχών. Ε, σας ευχαριστώ λοιπόν για την επικοδομητική υποστήριξη. Θα χρειαστούμε κι άλλοι στου επόμενους μήνες και ε, πρέπει... εκ παραλίλου να προσπαθήσουμε να πείσουμε και τις επιχειρήσεις να αλλάξουν προσέγγιση. Αυτά προς το παρόν από πλευράς μου και είμαι στη διάθεσή σας να συζητήσουμε. Ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Ευχαριστώ κυρία Επίτροπε για την παρουσίασή σας και τώρα θα αρχίσουμε τη συζήτηση. Θα αρχίσουμε με έναν πρώτο κύκλο ερωτήσεων με παρεμβάσεις από τους συντονιστές και θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Λεγκρίπ. Παρακαλώ. Oui, merci, euh, madame la... Ναι, σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ σήμερα. Θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω διότι κάνατε μια πολύ μεγάλη επισκόπηση στην ουσία που μας επιτρέπει να έχουμε πιο επίκαιρες πληροφορίες και να μπορέσουμε να συζητήσουμε και να δούμε τις μελλοντικές μας εργασίες, ε, την πιθανή κινητοποίηση που θα έχουμε στο μέλλον. Δύο ερωτήσεις έχω για το σχέδιο οδηγίες ε, για τις γυναίκες στα διοικητικά συμβούλια, το Women on Boards. Ε, μας είπατε βέβαια ε, κάποια πράγματα. Συμφωνώ με την απογοήτευσή σας και με την ανησυχία σας ε, και εξ ονόματος πολιτικής μου ομάδος ελπίζω ότι θα υπάρξουμε νεότερα. Ε, μπορείτε βεβαίως ε, να βασίζεστε στην πλήρη αποφασιστικότητά μας για το θέμα αυτό, όπως και για άλλα θέματα και σας ευχαριστούμε που ε, προσπαθήσατε ουσιαστικά να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες. Η ερώτησή μου αφορά την κατάσταση και την πρόοδο των εργασιών όσον αφορά την κύρωση της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης. Σας ευχαριστώ επίσης που μας δώσατε και τις πληροφορίες και επομένως θεωρούμε ότι στις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να οριστικοποιήσουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε να περάσουμε στην οριστική κύρωση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για άλλη μια φορά λοιπόν σας ευχαριστώ για όλες αυτές τις προσπάθειες. Ξέρουμε ότι η προσωπική σας πρωτοβουλία και η προσωπική σας δέσμευση ήταν πάρα πολύ μεγάλη και αποφασιστική σημασίας πιστεύω και η ομάδα του ΕΛΚ παρακολούθησε με ιδιαίτερη ε, αφοσίωση το θέμα αυτό. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο θέματα. Η Επιτροπή Γυναικών πριν από λίγο ενέκρινε ε, την έκθεσή μου για την ανάγκη να υπάρχει μια ευρωπαϊκή στρατηγική για τη μείωση των ανισοτήτων ε, στις συντάξεις. Το λεγόμενο Gender Gap in Pensions. Και να δούμε πώς θα πάει η ψηφοφορία στην Ολομέλεια στον Ιούνιο για αυτή την έκθεση που μόλις εγκρίθηκε. Ε, θα υπάρξουν αρκετές ευκαιρίες να το συζητήσουμε πρόσφατα και στην Ολομέλεια διότι θα γίνει συζήτηση και ψηφοφορία στην Ολομέλεια και θα ήθελα να σταθώ και σε κάτι συγκεκριμένο. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει πολύ συγκεκριμένη δουλειά και εις για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε ε, την κατάσταση και να έχουμε ε, αξιόπιστους δείκτες αποτελεσματικούς και σοβαρούς που θα μας επιτρέπουν να έχουμε την κατάλληλη μεθοδολογία για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε και να διευκρινίσουμε ε, την εικόνα της κατάστασης που έχουμε για τη διαφορά που υπάρχουν στις συντάξεις μεταξύ γυναικών, διότι η κατάσταση είναι σκανδαλώδης αυτή τη στιγμή. Βλέπουμε όμως ότι πρέπει να βελτιώσουμε την μέθοδό μας και να μπορέσουμε να έχουμε καλούς δείκτες και να μπορέσουμε να εργαστούμε και να φροντίσουμε ε, να μπορούμε να ε, προτείνουμε κάποια πράγματα από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη που να είναι αποτελεσματικά και τα κράτη-μέλη να βοηθηθούν ώστε να λάβουν τι κατάλληλε αποφάσει επειδή θα έχει γίνει κατάλληλη διάγνωση κατάσταση. Αναφερθήκατε στο πνεύμα τη δέσμη μέτρων για την ε, ισορροπία μεταξύ οικογενειακή και επαγγελματική ζωή και σε αυτό το σημείο ε, σημειώνουμε πώς δεσμευτήκατε προσωπικά για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Ε, δεν είναι και τόσο ερώτηση, διότι αυτή τη στιγμή τώρα αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τις λεπτομέρειες ε, των προτάσεών σας και τις ε, θέσεις σας, αλλά από πλευράς ΕΛΚ σας διαβεβαιώ ότι θα έχουμε μια πολύ δραστήρια και επικοδομητική στάση και θα προσπαθήσουμε να είμαστε επικοδομητικοί και θετικοί και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, αν μπορούμε να συμπληρώσουμε και να βελτιώσουμε, να είμαστε δύναμη στήριξη ε, σεβόμενοι και τις θέσεις των κρατών μελών, αλλά ταυτόχρονα και τις ε, κοινέ μας αξίες ε, και αρχές, για να μπορέσουμε να προωθήσουμε και την κοινωνική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που περιμένουν οι Ευρωπαίοι συμπατριώτες μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκαρσία Πέρες, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία ε, να ευχαριστήσω. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω την κυρία Γιούρεβα που ήρθε στην Επιτροπή μας. Εδώ και αρκετό καιρό περιμέναμε να έρθετε. Σας καλωσορίσουμε λοιπόν. Πιστεύω ότι στο χώρο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ακούσουμε τι ακριβώς κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα της αρμοδιότητές μας ε, και εσείς ε, ταυτόχρονα μπορείτε να μάθετε τις ε, βασικές ανησυχίες των μελών της Επιτροπής μας. Πιστεύω ότι κάνατε μία επισκόπηση για τα σημαντικά θέματα που μας απασχολούν αυτή τη στιγμή και θα είμαι πολύ σύντομη. Καταρχάς θα θέλαμε να καλωσορίσουμε την πρόταση για τη συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Την περιμέναμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και θεωρώ ότι έρχεται να απαντήσει σε μία από τις προσδοκίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δηλαδή να υπάρξουν συγκεκριμένες νομοθετικές προτάσεις. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η σε πολλές περιπτώσεις μόνο μέσω της νομοθεσίας μπορούμε να έχουμε τελικά μία δεσμευτική πολιτική για κάποια θέματα. Ελπίζω λοιπόν να έχουμε και εμείς τη δυνατότητα εδώ στο Κοινοβούλιο να συζητήσουμε, να βελτιώσουμε το κείμενο για τις γονικές άδειες, αλλά από πλευράς μου πιστεύω ότι αποτελεί μια πολύ καλή αρχική πρόταση, ένα πολύ καλό σημείο κίνησης το οποίο θα μπορέσουμε ελπίζω να βελτιώσουμε εδώ στο Κοινοβούλιο και επίση ελπίζω ότι δεν θα μα συμβεί τελικά αυτό που έγινε και με την οδηγία για την άδεια μητρότητα, δηλαδή να μπλοκάρει το θέμα στο Συμβούλιο. Ε, ελπίζω λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει φροντίσει να προσπαθήσει να πείσει τα κράτη-μέλη για τη σημασία που υπάρχει για να προχωρήσουμε στα θέματα συμφωλίωσης οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Υπάρχει και ένα θέμα το οποίο μας απασχολούσε όσον αφορά τη μητρότητα και τις απολύσεις, διότι ε, γνωρίζουμε κάποιες περιπτώσεις και μας είχατε πει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να αντανακλάτε κάπου αυτή η κατάσταση και λέτε ότι δεν έχουν τεθεί σε νομοθετικό επίπεδο, αλλά πρόκειται για μια ανταλλαγή καλών πρακτικών γιατί υπάρχει ήδη νομοθεσία από αυτού. Θα ήθελα να ξέρω αν έχετε κάποιες πληροφορίε εδώ, Αλλιώ μπορείτε να μα τι διαβιβάσετε σε κάποια άλλη στιγμή, ε, να τι στείλετε στα μέλη τη Επιτροπής Ποια συγκεκριμένη ε, νομοθεσία υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο όπου προστατεύεται η εργαζόμενη έγκυος γυναίκα, διότι θα ήθελα να μπορέσουμε να ελέγξουμε ότι όντως έγινε και τα κατάλληλη μεταφορά στην εθνική νομοθεσία. Διότι όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, η πραγματικότητα σήμερα είναι ότι δεν τηρείται η νομοθεσία. Υπάρχουν ακόμα γυναίκες στην Ευρώπη, εργαζόμενες, οι οποίες απολύονται απλώς και μόνο διότι ε, εγκυμονούν. Επομένως, ε, θα ήθελα να ξέρω ακριβώς ε, πού είναι η νομοθεσία που αναφέρει ε, τη συγκεκριμένη διάταξη και αν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς έγινε η μεταφορά της στα κράτη-μέλη. Και επίσης, και με αυτό ολοκληρώνω, αναφερθήκατε στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Κάνατε μια πολύ σημαντική προσπάθεια. Το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή μας επίσης έκανε μεγάλη προσπάθεια έγινε η συζήτηση για την ε, έμφυλη βία αρκετές φορές και στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η έμφυλη βία είναι ένα από τα πιο επωνίδιστα στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Επομένω, για μα η κύρωση τη Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη είναι θεμελιώδη σημασία. Αναφερθήκατε σε ένα συμβιβαστικό κείμενο και είπατε ότι ε, κατέληξε το Συμβούλιο σε συμβιβασμό και θα ήθελα να ξέρω αν μπορείτε να μα δώσετε κάποιε περαιτέρω πληροφορίε από αυτού εάν αυτό το συμβιβαστικό κείμενο ε, σημαίνει ότι κυρώνεται το σύνολο της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ή γίνεται επιλογή κάποιων θεμάτων τα οποία θεωρούνται από πλευράς ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι είναι ε, νομοθεσία που αφορά τα θέματα αυτά μας. Δηλαδή, θα υπάρξει πλήρω κύρωση τη σύμβαση τη Κωνσταντινούπολη βάσει αυτού του συμβιβαστικού κειμένου ή θα κυρωθούν μόνο κάποια τμήματα τη σύμβαση. Αν μπορείτε να μα απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση και επίση θα ήθελα, εάν δεν μπορείτε, να μα στείλετε πληροφορίε ε, όποτε θεωρείτε εσεί ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Σα ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σα εδώ σήμερα. Thank you and... Ευχαριστώ. Thank you very much, uh, Madam Chair. Thank... Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τον χρόνο που διαθέσατε για να μας δώσετε τις λεπτομερίες αυτές τις πληροφορίες. Το εκτιμούμε πάρα πολύ. Ήδη το είπαν και οι συνάδελφοι. Θα ήθελα να σας πω πως η ομάδα του Άλντε επικροτεί τις προτάσεις που κάνατε. Τις θεωρούμε ως σύγχρονες κατάλληλες για τον 21ο αιώνα. Πιστεύουμε πως τα εργαλεία αυτά θα βοηθήσουν για την βελτίωση της απασχολησιμότητας των γυναικών και όπως είπατε, αυτό είναι κάτι που θα υποφελήσει την οικονομία. Στο σύνολό της έχει το δυναμικό να αυξήσει τα έσοδα και να προκαλέσει καλύτερη επαγγελματική ανέλυξη και έτσι θα έχουμε με τις γυναίκες στην αγορά εργασία μια μεγαλύτερη δεξαμενή δεξιοτήτων. Οι ελλείψεις θα πρέπει να αντιμετωπιστούν και έτσι θα μπορέσει να υπάρξει καλύτερη προσέλκυση εργαζομένων, θα υπάρχουν καλύτερα κίνητρα για τους εργαζόμενους. Οπότε αυτό θα έχει θετικές επιπτώσεις για την παραγωγικότητα των επιχείρησεων και αυτό θεωρούμε εμείς πως είναι ο κατάλληλος Πώς να επιτευχθούν όλα αυτά. Υποστηρίζουμε τις νομοθετικέ και τις μη νομοθετικές δράσεις. Θα έλεγα λοιπόν πως πρόκειται για μια δέσμη μέτρων η οποία είναι καλή και όπως είπατε δεν πρόκειται μόνο για νομοθεσία αλλά για μια συνεκτική πολιτική το οποίο το καθιστά ενδιαφέρον για μας όσον αφορά το σχόλιο σας για τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Ήδη κάποιοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν σε αυτήν. Θα ήθελα να σχολιάσω ξεκάθαρα την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών ως εργαλείο κατά της βίας κατά των γυναικών. Και πιστεύω ειλικρινά πως αυτό το έχω πει πολλές φορές, θα το επαναλάβω και μια φορά σε αυτό το πλαίσιο. Η οικονομική εξάρτηση είναι επικίνδυνη για τη ζωή και πρέπει να την υπερβούμε. Αυτό που είπατε, Επίτροπε, επίσης ξεκάθαρα, είναι πως η βία κατά των γυναικών γίνεται ακόμα ευρέως αποδεκτή στις κοινωνίες μας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συνεχιστεί. Τέλος, ένα γενικότερο σχόλιο, περισσότερο για τους συναδέλφους μου εδώ. Θα ήθελα να τονίσω την πρόταση της Άλντε για τα σεξουαλικά δικαιώματα καλούμε την Επιτροπή να προωθήσει τα δικαιώματα αναπαραγωγής και τα σεξουαλικά δικαιώματα την επόμενη περίοδο. Ακόμη οι ομάδες μπορούν να προσθέσουν στοιχεία. Η ψηφοφορία θα γίνει στις 11 Μαΐου εδώ στην Επιτροπή ΦΑΜ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν θα θέλατε ίσως να σχολιάσετε ή να υποστηρίξετε το κείμενο αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ η κυρία Μπιόρκ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Επιτροπό Γιούροβα για την προσέλευσή της εδώ. Λίγα μονολόγια για το πολύ σημαντικό πακέτο για το συνδυασμό επαγγελματική και ιδιωτική ζωή. Είναι πολύ θετικό που επιτέλου μια δέσμη μέτρων που εστιάζει όντω στον πυρήνα τη συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασία κατατίθεται ξανά Υπάρχουν στοιχεία που είναι εξαιρετικά σημαντικά όπως είναι η μη δυνατότητα μεταφοράς, transferability, όπως είναι οι αμοιβέ, οι επιλογές για άντρες και τους γυναίκες. Θα ασχοληθούμε και θα συζητήσουμε και εδώ για ευέλικτες σχέσεις εργασίας ως γενική ρήτρα Πιστεύω πως πρέπει να ασχοληθούμε με το, με το ζήτημα αυτό επίσης. Επίσης, πιστεύω πως μέσω των μη νομοθετικών μέτρων μπορούμε να επενδύσουμε στην υποδομή για την φροντίδα των παιδιών. Το ένα δεν θα λειτουργούσε χωρίς το άλλο, αλλά έχουμε δυνατότητα να επανέλθουμε στη δεσμή μέτρων αυτή και να εργαστούμε επ' αυτή στην Επιτροπή αυτή, συνεργαζόμενοι και με εσάς, ώστε να γίνει όσο δυνατόν καλύτερη. Δύο πράγματα μόνο ακόμα που θα θέλω να θέσω Πιστεύω πως είναι πολύ απαιτητικό για εσάς ως αρμόδιας επιτρόπου. Έχει τεθεί στην Επιτροπή. Είναι ο κανόνας της ολικής φήμωσης που απειλεί τα σεξουαλικά και αναπαραγωγικά δικαιώματα των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Και εσείς ως αρμόδια επίτροπος θα πρέπει σε συνεργασία και με τους άλλους επιτρόπους αλλά και με τη δική μας υποστήριξη θα πρέπει να υποστηρίξετε με πολύ ενεργό τρόπο την ελευθερία των γυναικών σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης θα ήθελα να θέσω το εξή. Ζητήσαμε από το Κοινοβούλιο για μια καινούργια στρατηγική κατά της εμπορίας ανθρώπων και στην Επιτροπή αυτή ήμασταν πολύ σαφείς ότι η εμπορία γυναικών και κοριτσιών για σεξουαλική εκμετάλλευση είναι το πιο σοβαρό ζήτημα. Χρειαζόμαστε μια πολύ ισχυρότερη προοπτική της συνεκτίμησης της διάστασης του φύλου και όσον αφορά την σεξουαλική εκμετάλλευση. Καμία στρατηγική ενάντια στην εμπορία ανθρώπων δεν θα είναι επιτυχής χωρίς αυτό. Έθεσα στον Επίτροπο Αβραμόπουλο την ερώτηση αυτή, αλλά πιστεύω πως είναι η δική σας τεχνογνωσία που χρειάζεται εδώ. Ένα ακόμα και τελειώνω. Μπορεί να μην απευθύνεται άμεσα σε εσά, αλλά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάσισε πως ο εργοδότης έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσληψη μιας υπαλλήλου εάν φοράει μαντήλα. Πιστεύω πως αυτό ανοίγει τις πόρτες για τις διακρίσεις εις βάρος των γυναικών στην Ευρώπη και πιστεύω πως αυτή δεν είναι μια αποδεκτή εξέλιξη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με τέτοιες εξέλιξεις στη σημερινή Ευρώπη. Και πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά πώ να μην ανοίξουμε τι πόρτε αυτέ προ τι διακρίσει. Χρειαζόμαστε όλε τι γυναίκε στην αγορά εργασία και όχι μόνο κάποιε. Ζητώ συγγνώμη επειδή έχω υποχρέωση σε μια άλλη επιτροπή, αλλά συνάδελφοί μου βρίσκονται εδώ και εγώ θα συνεργαστώ ευχαρίστω όπω και αυτή μαζί σα, Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ο κ. Μαξελέ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και την κυρία Γιούροβα για τη σημερινή της παρουσία εδώ από πλευράς ε, Ευρωπαίων Πρασίνων ε, καλωσορίζουμε αυτή την πρόταση για τη συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Πιστεύουμε ότι ε, προτείνει θετικά μέτρα, όπως για παράδειγμα τις, τους τέσσερις μήνες γονικής άδειας και είναι βελτίωση. Ξέρετε βεβαίως ότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι στο 100%. Ε, φαίνεται ότι έχουμε υποχωρήσει στις φιλοδοξίες μας, ιδίως σε σχέση με την οδηγία για την άδεια ε, διότι εξακολουθούν να απουσιάζουν πολλά στοιχεία ε, σε αυτά τα οποία παρουσιάστηκαν. Βέβαια, ε, γνωρίζοντας και την αντίθεση του Συμβουλίου, είναι πολύ σημαντικό αυτό και επίσης ε, ε, ελπίζουμε επιτέλους να γίνει υποχρεωτική γονική άδεια και να είναι αμοιβόμενη. Το λέω γιατί φαίνεται ότι είμαι ο μόνος άντρας. Υπάρχουν και πατέρες λοιπόν και οι πατεράδες μπορούν να βοηθήσουν στη συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου και επομένω γι' αυτό πρέπει να δώσουμε περισσότερα δικαιώματα στους άντρες για να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε και εμείς στον οικογενειακό βίο και να φροντίσουν και οι γυναίκες να έχουν περισσότερα δικαιώματα με τη σειρά τους. Θα ήθελα να σταθώ στα μη νομοθετικά μέτρα, κυρίως ένα στοιχείο κλειδί το οποίο πιστεύω ότι δεν σχολιάστηκε παρκώς, το θέμα της εποπτείας, της εποπτείας και της παρακολούθησης των μέτρων αυτών των μη νομοθετικών. Θα ήθελα να ξέρω τι άποψη έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι σκοπεύει να κάνει για να παρακολουθήσει τα μη νομοθετικά μέτρα και την εφαρμογή τους, ε, ιδίως ε, σε σχέση με τα Ευρωπαϊκά Περιφερειακά Ταμεία, στα κράτη-μέλη για τη βελτίωση των υποδομών, ε, για παράδειγμα, για... Ε, φροντίδα παιδιών, ε, βρεφονιπιακού ε, σταθμούς, νηπιαγωγεία κλπ. Και τι σκοπεύετε να κάνετε για να προχωρήσει αυτή η επικοινωνία, ε, διότι ξέρω ότι στο διάλογο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου έχετε υπόψη σας να συμπεριλάβετε και όλα αυτά τα θέματα, αλλά θα ήθελα να ξέρω πώς σκοπεύετε να έχετε και μια παρακολούθηση που θα επιτρέψει να υπάρξει αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των μη νομοθετικών μέτρων. Επίσης, θα ήθελα να σχολιάσω και κάτι ακόμα το οποίο δεν αναφέρατε εσεί στην παρέμβασή σας, αλλά θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, λαμβάνοντας υπόψη και το πώ ζούμε ε, ε, την κλιματική αλλαγή. Γνωρίζετε ότι εμείς από πλευράς Επιτροπής μας ξεκινήσαμε μια πολύ σημαντική δουλειά για την ε, κλιματική δικαιοσύνη με έμφαση στα θέματα φύλου. Και επειδή εσεί είστε υπεύθυνοι για την ισότητα των φύλων, θα ήθελα να ξέρω πώ βλέπετε τα θέματα αυτά τη κλιματική. Δικαιοσύνη. δικαιοσύνης ε, και ε, ε, τι κάνει η Γενική σας Διεύθυνση για τα θέματα αυτά. Ασχολείστε με τα θέματα κλιματικής δικαιοσύνης και αν συνεργάζεστε και με τον Αρμόδιο Επίτροπο για τα θέματα κλίματος, διότι το θέμα της κλιματικής δικαιοσύνης είναι ένα οριζόντιο ζήτημα το οποίο έχει σχέση και με τον Επίτροπο αλλά και με την Επίτροπο Δικαιοσύνης και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια πολύ σημαντική δέσμη μέτρων, ε, τα λεγόμενα μέτρα του χειμώνα, η καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους. Πρέπει να υπάρχει και σαφής αναφορά στη διάσταση του φύλου σε αυτά τη δέσμη μέτρων για το χειμώνα, εάν θέλουμε η ενεργειακή απόδοση να έχει στο επίκεντρο τις γυναίκες ε, στις δράσεις αυτές. Και θα ήθελα να ξέρω εάν προτείνατε στον πρόεδρο Γιούγκερ, για παράδειγμα, κάτι σχετικό και αν ζητήσατε το δικό σας το γραφείο να συμμετέχει και στην δέσμη μέτρων για το κλίμα. Εάν δηλαδή το θέμα του φύλου ε, περιλαμβάνεται και στα θέματα της ενεργειακής μετάβασης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω α, το λόγο ε, στην Επιτροπή του ώστε να δώσει κάποιες απαντήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για τα ερωτήματα και τα σχόλιά σας. Ε, κάποια έμπνευση την οποία μου δώσατε. Πρόεδρε, με, με σύντομο τους ώστε να θέσουν περαιτέρω ερωτήματα μέλη της Επιτροπής. Πρόεδρος, ε, ναι, ε, καλά, καλά θα ήταν να μην τώρα ώστε να δεθούν περαιτέρω ερωτήματα. Επιτροπός. Καλώς θα ε, μας Οπότε... θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχήν και προσωπικά για το, για το ενδιαφέρον σας και για το γεγονό ε, ότι εκτιμάτε τις προτάσεις ε, του πακέτου για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ε, ζωής, κυρία Λεκρύπα, αλλά εντάξει, όταν σκεφτόμαστε βέβαια αυτό το καθεστώς θα πρέπει να σκεφτόμαστε και το τι συμβάνει και με εμάς τους ίδιους, αλλά Νομίζω πως ε, έχουμε ακόμα κάποιες ε, ελπίδες αφού βρίσκομαστε στην αρχή. Ίσως δηλαδή θα μπορέσουμε να ε, συνδυάσουμε καλύτερα τις υποχρεώσεις που έχουμε, δηλαδή και εμείς οι ίδιοι, οικογενειακές και επαγγελματικέ. Τώρα, θα πρέπει να εργαστούμε έτσι ώστε αυτή η ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτική ζωή να αποτελέσει ένα από τα βασικά εργαλεία για την αντιμετώπιση τη μισθολογική ανισότητα και κατά συνέπεια και τη συνταξιοδοτική ε, ε, ανισότητα. Ε, σε κάποια κράτη-μέλη αυτή μπορεί να είναι πολύ ψηλή, να φτάνει στο 30%, σε κάποια μέρη και στο 40%. Είναι πραγματικά ανησυχητική η κατάσταση και διαπιστώνουμε ότι η κύρια πηγή αυτής σύνταξη ανισότητας είναι, είναι ε, φροντίδα των εξαρτώμενων μελών της από, την, ε, από τη γυναίκα μέσα στην οικογένεια. Έτσι λοιπόν προσπαθούμε να λάβουμε υπόψη μας ακριβώς αυτή τη φροντίδα που προσφέρουν οι γυναίκες στα μέλη της οικογένειάς τους. Οπότε ε, πρέπει εδώ να αναφέρουμε ξεκάθαρα το τι συμβαίνει. Και να αποδίδουμε τις ευθύνες γιατί πραγματικά δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η ανισότητα και ε, συμφωνώ πλήρως μαζί σας ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε σε μια ανάλυση και ε, στην ανάπτυξη μια σειράς ε, αποτελεσματικών δικτών, τόσο ώστε να μπορούμε να μετρούμε αυτό το φαινόμενο. Εγώ στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ θα προτείνω στους υπουργού, το πιθανότερο στο Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ του Ιουλίου από την Εστονική Προεδρία, κάτι σχετικό. Γιατί ζήτησα από αυτή την Προεδρία να συμπεριλάβει το ζήτημα της συνταξιδοτικής ανισότητας στα ε, σημεία προσυζήτηση ε, του εν λόγω Συμβουλίου το ταχύτερο δυνατό. Και αυτό γιατί, γιατί η Επιτροπή μέσα στο δεύτερο εξάμεινο του 2017 θα προτείνει το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος της μισθολογικής ανισότητας και σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα της συνταξιοδοτικής ανισότητας. Οπότε ε, ειδικότερα οι Υπουργοί Εργασία και Κοινωνικών Υποθέσεων αποτελούν ένα πολύ σημαντικό φόρουμ ούτω ώστε να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο ε, τη μισθολογική ανισότητα, δηλαδή το τι συμβαίνει κατά την ε, επαγγελματική σταδιοδρομία των γενικών, αλλά και το τι συμβαίνει σε επίπεδο του ανισότητα. Στο πλαίσιο τώρα αυτού του σχεδίου δράση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλε τι αιτίε που οδηγούν σε αυτήν την ανισότητα και οι οικογενειακές υποχρεώσεις αποτελούν μια πολύ σημαντική πηγή όπω είπα. Μια ε, άλλη ε, πηγή είναι οι δυσμενές ε, διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, δηλαδή διαφορετικές αμοιβέ για την ίδια εργασία. Πράγμα το οποίο προφανώς αποτελεί μία ευθύνη των αρχών εποπτείας της αγοράς εργασίας, δηλαδή των αρχών εκείνων που είναι υπεύθυνε για την επιβολή του νόμου, έτσι ώστε να προσφέρουν υποστήριξη στα θύματα μιας τέτοιας, ε, τέτοιων δυσμενών ε, διακρίσεων, ώστε να ε, υπάρξει την κατάλληλη προσφυγή. Γιατί βλέπουμε συχνά ότι τα θύματα μια τέτοια δυσμενού μεταχείριση στην εργασία του συχνά δεν έχουν δυνατότητες να λάβουν υποστήριξη σε κοινωνικό επίπεδο. Δηλαδή τα θεσμικά όργανα δεν τους προσφέρουν αυτή την υποστήριξη και αυτό θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Έτσι λοιπόν θα πρέπει εδώ να εμπλέξουμε πιο ενεργά τις αρχές εποπτείας της ε, αγοράς εργασίας, πράγμα το οποίο ήδη ε, κάναμε στο πλαίσιο του πακέτου για το Work Life. Ε, τώρα, μία ακόμα αιτία η οποία οδηγεί στην, σε αυτή την μισολογική και κατά συνέπεια σε ταξιδιωτική ανισότητα είναι η, τα διαχωρισμένα, αν θέλετε, παντήματα. Και εδώ ουσιαστικά πρόκειται για το δυσκολότερο ζήτημα, γιατί μόλις ένα συγκεκριμένο επάγγελμα θεωρηθεί γυναικείο εντό εισαγωγικών επάγγελμα, αυτομάτω ε, αυτό συνεπάγεται χαμηλότερη αμέμενη. Και αυτό ε, δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη έκπληξη όταν διαπιστώσουμε ότι ισχύει κυρίως στο δημόσιο τομέα των κρατομελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν μέσω συστάσεων ανά κράτος μέλος, εξετάζοντας δηλαδή την κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος, είναι η καταλληλότερη ε, πρόταση και από εκεί και μετά θα δούμε πώς μπορούμε να προτείνουμε περαιτέρω λύσεις για την αντιμετώπιση της ε, μισθολογικής ανισότητας. Εάν έχετε κάποιες ιδέες από την πλευρά σας σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, ε, για αυτά τα επαγγέλματα, αν θέλετε, τα οποία έχουν θεωρούνται ότι ανήκουν σε ένα από τα δύο φύλλα. Θα ήθελα να τις ακούσω γιατί δεν θέλουμε απλά να θέσουμε μια ποσόστοση σε ό,τι αφορά την εκπροσώπηση των ανδρών σε αυτά τα επαγγέλματα. Εντάξει, αστείευομαι, αλλά ε, από εκεί και μετά ένα ακόμα πρόβλημα ε, σε ό,τι αφορά αυτή την ανισότητα είναι το γεγονός ότι οι ανάκοριστα και οι γυναίκες, οι νέες γυναίκες δεν επιλέγουν τις σπουδέ εκείνες οι οποίες οδηγούν σε καλύτερα αμοιβόμενα επαγγέλματα. Για παράδειγμα, ο τομέας της πληροφορικής Χρειάζεται επιγόντως νέα ταλέντα, νέες γυναίκες που έχουν έναν διαφορετικό τρόπο σκέψης, ε, και φέρνουν καινοτομίε. Και μα λέει αυτό ο κλάδο ότι οι γυναίκε δεν συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, ακριβώ δεν έχουν επιλέξει τι κατάλληλε σχολέ και δεν έχουν επιλέξει τι κατάλληλε σπουδέ προ αυτή την κατεύθυνση. Οπότε λοιπόν έχουμε συμπεριλάβει ε, στην δική μα ατζέντα για τι δεξιότητε ε, των συνάδελφων επιτρόπων ένα στοιχείο το οποίο ακριβώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη καλύτερη επιλογής των αντικειμένων σπουδών, μεταξύ δηλαδή αρών ανδρών και γυναικών. Αυτό λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε με διαφορετικές έλευσεις. Και από εκεί και μετά, ένα περαιτέρω ε, λόγο για αυτή την ανισότητα είναι η χαμελή αυτοπεποίθηση των γυναικών. Δηλαδή δεν αξιώνουν καλύτερε αμοιβέ. Όπου δηλαδή πηγαίνω εγώ και συναντώ ε, και τι γυναίκε, αυτό τους λέω. Δηλαδή αξιώστε την κατάλληλη αμοιβή για το επάγγελμά σα. Δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι κανείς ε, επιφυλακτικός, διστακτικός. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να αναπτύξουμε εδώ όχι μια στρατηγική αλλά ένα έγγραφο το οποίο θα εκθέτει όλα αυτά τα προβλήματα, ε, τις πηγές δηλαδή οι οποίες οδηγούν τελικά, τις αιτίες ε, οι οποίες οδηγούν στην ανισότητα και θέλουμε ε, ε, να επιτύχουμε καλύτερη, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη δικαιοσύνη, περισσότερες ε, συστάσεις ανακράτος μέλος, καλύτερη ενσωμάτωση μέσα στην ατζέντα για τις δεξιότητες, εφαρμογή του πακέτου Work-Life Balance και ενδεχομένως αναθεώρηση της οδηγίας 2654 Γιατί ίσως υπάρχουν κάποια κενά στην νομοθεσία τη σήμερα ημέρα, τα οποία ενδεχομένω με μια αναθεώρηση τη εν λόγω οδηγία ε, μπορούν να αντιμετωπιστούν. Αυτέ είναι οι αρχέ μα προτάσει, ώστε να υπάρξει περισσότερη διαφάνεια τόσο στο επίπεδο τη αναθεωρημένη νομοθεσία, αλλά και στο επίπεδο των, επιβολή επιβολής ε, κυρώσεων. Σε ό,τι αφορά δηλαδή την εφαρμογή τέτοιων πρακτικών ε, διακρίσεων ε, στους, ε, στην εργασία. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά το γενικότερο σχέδιο δράση μα και αναμένω βέβαια με ενδιαφέρον τι δικέ σα προτάσει, γιατί εσεί βρίσκετε σε συνεχή επαφή με του δικού σα ψηφοφόρου και έχετε πολλά πρακτικά παραδείγματα τα οποία μπορείτε να μα αναφέρετε. Νομίζω πως κάλυψα τα σχόλια που έγιναν ε, σε ό,τι αφορά την ε, ισορροπία μεταξύ οικογενειακή και ιδιωτικής ζωής. Τώρα, ε, τις ελπίδες μας ε, ε, Ω προ το αυτά θα γίνουν δεκτά από το Συμβούλιο ή όχι, αυτά που μα είπε δηλαδή ε, κυρία Γκαρσία Περεσέ. Είχαμε μια κακή εμπειρία όπω σα είπα με την οδηγία σε ό,τι αφορά την ε, άδεια μητρότητα. ε, και το Συμβούλιο τι μα είπε εκεί ουσιαστικά μα μπλόκαρε και μα είπε ξαναρχίστε από την αρχή και κάντε μια καλύτερη πρόταση. Εμεί νομίζουμε πω δεν θα υπάρξει μια αυστηρά αρνητική αντίδραση από την πλευρά του Συμβουλίου. Έχουμε συζητήσει δηλαδή το αν λόγω ζήτημα επανειλημμένα με του ε, υπουργού, αλλά τον Ιούνιο θα γίνει για πρώτη φορά συζήτηση συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά αυτό το πακέτο προτάσεων. Και αυτό που εμεί ακούμε ήδη ότι θεωρείται προβληματικό από το Συμβούλιο ε, σε ό,τι αφορά το νομοθετικό τμήμα είναι το ζήτημα της χρηματοδότησης ότι δηλαδή η γονική άδεια θα πρέπει να λαμβάνει αποδοχές, να αποζημιώνεται με αποδοχές αντίστοιχες με αυτές τις άδεια ασθενείας. Ε, εντάξει, εμείς ε, ε, δεν μπορούμε να είμαστε αρμόδιοι για το ποιος θα κληθεί να καταβάλει τέτοιου είδους επιδόματα αδείας, κατά πόσο δηλαδή εργοδότες θα κληθούν να το πράξουν ή τα ταμεία κοινωνική εκείνο που εμείς έχουμε είναι μακροοικονομικά στοιχεία, πολύ πιστικά και συγκεκριμένα στοιχεία όπου ε, βράχει πρόθεσμα, οι δαπάνες ενδεχομένως θα αυξηθούν λίγο, αλλά μακροπρόθεσμα τα ωφέλη θα είναι πολύ ισχυρά. Και αυτά τα επιχείρηματα θα εκθέσουμε στο πλαίσιο του διαλόγου που θα κάνουμε με τα κράτη-μέλη. Όταν θα ακούσουμε δηλαδή ακριβώς αυτά τα αντεπιχειρήματα από την πλευρά τους που μόλις σας εξέθεσα. Τώρα, σε ό,τι αφορά την προστασία των τέρων και γενικότερα των γονέων, ήδη υπάρχει ε, στην οδηγία ε, για την ε, γονική άδεια η απαγόρευση της, της μενούς διάκρισης σε ό,τι αφορά ειδικότερα ε, τις ε, απολύσεις και εδώ μιλάμε δηλαδή για μια νομοθεσία η οποία πρέπει να εφαρμόζεται. Και αυτό το είπα όταν σας ανέφερα εισαγωγικά το πακέτο για την ισορροπία μεταξύ επαγγελματική και ιδιωτικής ζωής. Δηλαδή η επιβολή αυτής της νομοθεσίας θα πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματικά και θα πρέπει ταυτόχρονα να αυξηθεί και η εμπιστοσύνη των ε, μητέρων, των πατέρων και των φροντιστών τι ε, αρμόδιες αρχές υποστηριξή του, ώστε να μπορούν να επεμβαίνουν και να επιλύουν τις ε, εν λόγω διαφορές. Άρα λοιπόν αυτή η προστασία ήδη περιλαμβάνεται στην υφιστάμενη νομοθεσία, αλλά και στη σχετική οδηγία που προτείνουμε τώρα στο άρθρο 12 υπάρχει προστασία από απόλυση για όσους εχαίρουν των σχετικών δικαιωμάτων ε, ε συμπεριλαμβανομένες της ε, και άδεια φροντιστών προσπαθούμε ακριβώς εδώ να ενισχύσουμε την προστασία των γονέων και των ε, φροντιστών μέσω της συμπερίληψης του άρθρου 12, προστασίας πάντα από ε, απολύσεις. Στο 12 Και από εκεί και μετά υπάρχει και η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση Ντέκερ, όπου καθίσταται απόλυτα σαφές ότι υπάρχει ανάγκη να εφαρμόζεται στο ακέραιο η προστασία ε, των φροντιστών ε, των ε, μητέρων και των γονέων γενικότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, μπορώ να σας παράσχω γραπτές απαντήσεις, γιατί πρόκειται για μια περίπλοκη νομική υπόθεση, αλλά εν συντομία μπορώ να σας απαντήσω τώρα. Πω το εξής. Εμείς προσπαθούμε να προτείνουμε ε, το μεγαλύτερο δυνατό ε, ή το ευρύτερο δυνατό φάσμα αρμοδιοτήτων για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η τελική εκδοχή αυτής της σημασίας μάλλον θα ε, περιορίσει τις αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ναι. επιτρέψει δηλαδή μόνο εκείνες τις αρμοδιότητες τη Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι αποκλειστικές αρμοδιότητες τη και όχι μεικτέ με τα κράτη-μέλη. Ε, και αυτό πολύ σύντομα, όμω μπορώ να σα δώσω και γραπτές ε, απαντήσεις, γραπτά σχόλια ώστε να σας εκθέσω όλη τη διαδικασία που ακολουθήθηκε. Την στιγμή έχουμε ε, το συμβαστικό κείμενο σε ό,τι αφορά τι αποφάσει του Συμβουλίου, σε ό,τι αφορά την ε, υπογραφή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης ε, από την, ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχοντας λάβει τη σύμφωνη γνώμη της Κορεπέρ και μόνο η Πολωνία εδώ έχει επαναλάβει την αρνητική της θέση. Χωρίς, και από εκεί και μετά η Γερμανία, η Σουηδία, η Ιρλανδία και η Ελλάδα χωρίς να απορρίπτουν την υπογραφή προτείνουν κάποιες τροποποιήσεις σε ό,τι αφορά την υπογραφή και το τι ακριβώς αυτή θα σημαίνει της σύμβασης. Η Επιτροπή τώρα, όπως σας είπα, εξέφρασε τη λύπη της σε ό,τι αφορά ε, το περιορισμένο ε, ε, φάσμα, σε ό,τι αφορά τις σχετικές αποφάσεις. Πράγμα δηλαδή το οποίο δεν θα επιτρέψει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει σε όλα αυτά τα τμήματα τη Ανλογοσύμβαση σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα και εκφράζουμε επίση την ανησυχία μα σε ό,τι αφορά το κατακαιρματισμένο χαρακτήρα τη υπογραφή των αποφάσεων. Ε, αυτά θα τα αναφέρει και επισήμως ε, σε μια δήλωσή της και θα διαβιβαστούν στο Συμβούλιο ε, σχετικέ συστάσει προ Δεν γνωρίζουμε δηλαδή ακόμα ποια άκουσα θα επιλέξει το Συμβούλιο. Ο στόχος μας είναι όμως να συμφωνήσουμε το ταχύτερο δυνατό με το Συμβούλιο στις 11 Μαΐου. είναι μάλλον ε, περίπλοκη και η νομική βάση που έχει επιλεγεί για την ε, υπογραφή τη ε, Σύμβαση τη Κωνσταντινούπολης. Δηλαδή βρισκόμαστε στο το πεδίο της ποινική δικαιοσύνη και η νομική βάση είναι το 82 και το άρθρο 84 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά σε ό,τι αφορά τη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης. Κυρία πολύ ευχαρίστω να σας βοηθήσω για τον κύριο Μίμητσα. Για τη βία κατά των γυναικών, προφανώς και η οικονομική εξάρτηση είναι επικίνδυνη και υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία τα οποία καταδεικνύουν ότι αν δεν βοηθήσουμε τις γυναίκες να είναι πιο ανεξάρτητες ε, από οικονομική σκοπιάς, αν δεν τις βοηθήσουμε να έχουν καλύτερες αμοιβέ και να είναι λιγότερο ευάλωτε πάντα θα υπάρχουν υψηλά ποσοστά ε, ε, βίας, ε, κυρίως οικογενειακής βίας. Όλα αυτά είναι αλληλένθετα. Για τόσα είπε η κυρία Μπιόρκ, για την ευελιξία στη δέσμη μέτρων ε, για τη συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, προσπαθήσαμε πολύ σκληρά να μην κάνουμε λάθος στον τρόπο με τον οποίο θα ορίσουμε τη δυνατότητα ε, πιο ευέλικτων ε, ωραρίων για τις γυναίκες. Η κυρία Μπιόρκ αναφέθηκε σε μια πιθανή παγίδα και εμείς δεν θέλαμε να πέσουν οι γυναίκες σε αυτή την παγίδα. Η παγίδα θα μπορούσε να είναι η χρήση, ε, η εκμετάλλευση μάλλον της μερικής απασχόλησης. Αυτή είναι ε, χαρακτηριστική περίπτωση όταν οι γυναίκες προσπαθούν να συμφιλιώσουν ε, τα οικογενειακά τους καθήκοντα με τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, πέφτουν σε αυτή την παγίδα. Και τελικά χρειάζεται να δουλεύουν όσο σκληρά θα δούλευαν και αν ήταν πλήρως απασχολούμενοι, αλλά λαμβάνουν μισθό μερικής απασχόλησης. Ε, και κάνω μία απλή σύγκριση και προσπάθησα να δω τι σχέση υπάρχει μεταξύ του ποσοστού απασχόλησης γυναικών και ε, του μισθολογικού χάσματος. Και σε αρκετά κρατημέλη διαπιστώνουμε ένα πολύ περίεργο φαινόμενο. Όσο περισσότερο εργάζονται οι γυναίκες, τόσο μεγαλύτερο είναι το μισθολογικό χάσμα. Προσπάθησα να διαπιστώσω λοιπόν γιατί και το πρόβλημα βρισκόταν σε αυτές τις θέσεις δίθεν μερικής απασχόλησης, διότι ε, είναι ε, ε, μέτρα τα οποία θέτουν τις γυναίκες σε πολύ μειονεκτική θέση, γι' αυτό ακριβώς και δεν θέλαμε να πέσουν οι γυναίκες σε αυτή την παγίδα και σε άλλες παγίδες, πιέζοντας πολύ ε, σκληρά για αυτές τις δυνατότητες πιο ευέλικτων ωραρίων. Αυτό λοιπόν το, στο οποίο καταλήξαμε στην πρόταση είναι ότι εργαζόμενοι γονείς και άτομα που φροντίζουν άλλους μπορούν να ζητήσουν ευέλικτο ωράριο εργασίας ε, το οποίο προσφέρεται ανάλογα με τη μορφή και τη φύση της εργασίας αλλά ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να ε, εξετάσει το σχετικό αίτημα και να απαντήσει επί του αιτήματο. Και επίσης συμπεριλαμβάνουμε και ισχυρότερη προστασία για εκείνους που θέλουν να περάσουν και πάλι από μερική απασχόληση σε πλήρη απασχόληση, να μην υπάρχουν προσκόμματα στην αλλαγή αυτή. Επομένως, ε, ε, το εξετάσαμε αυτό πάρα πολύ προσεκτικά, ώστε να μην πέσουν οι γυναίκες στην παγίδα και να μην ε, καταλήξουμε σε κάποιο κοινωνικό σχεδιασμό το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες παρενέργειες. Το προσπαθήσαμε να τα εξισορροπήσουμε πάρα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Ε, καταπολέμηση του τράφικινγκ, αυτό είναι θέμα για τον Επίτροπο Βραμόπουλο, Σας απάντησε στις 3 Απριλίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το μόνο που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι συνεργαζόμαστε πάρα πολύ στενά με τον Δημήτρη Βραμόπουλο για ε, τα κοινά μα θεματολόγια Προσπαθώ να τονίσω την ανάγκη να έχουμε περισσότερη προστασία για ευάλωτους ανθρώπους, ιδιαίτερα γυναίκες και παιδιά, και στο θεματολόγιο ασφαλείας αλλά και στο θεματολόγιο για τη μετανάστευση. Όταν λοιπόν ε, ε, βλέπουμε τους κανόνες ασύλου και τους κανόνες του διβλούνιου θα δείτε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα τα οποία είναι αφιερωμένα σε ε, καλύτερη προστασία η οποία εγγυάται πλέον από την νομοθεσία για γυναίκες και παιδιά οι οποίοι ε, είναι μετανάστες. Για την εμπορία ανθρώπων υπάρχει η στρατηγική 2012-2016 ε, και τώρα βάσει και πληροφοριών από τον συνάδελφο τον κύριο Αβραμόπουλο εκπονούν τη νέα στρατηγική για το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και όλων των ενδιαφερομένων φορέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, υπάρχει ε, συγκεκριμένη διαβούλευση η οποία έγινε στο πρώτο εξάμεινο του 2016 με τα κράτη-μέλη, ε, με τους εθνικούς εισηγητές ή με αντίστοιχους μηχανισμούς, με υπηρεσίες δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων, πλατφόρμες της κοινωνίας των πολιτών για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Οι διαβουλεύσεις έγιναν και με διεθνείς οργανώσεις και με ομάδες της διοργανικής ομάδας ε, για την εμπορία ανθρώπων. Το νέο πλαίσιο πολιτικής θα έρθει να συγκεράσει όλους τους διάφορους αυτούς τομείς πολιτικής. Αυτά λοιπόν είναι ε, στη διαδικασία της εκπόνησης. Οι συνάδελφοι λοιπόν της κυρίας Μπιόρκ μπορούν να την ενημερώσουν ότι αν επιθυμεί περαιτέρω πληροφορίες μπορώ κάλλιστα να της δώσω ε, ό,τι θα μου δώσει ο κύριος Αβραμόπουλος. για την απόφαση του δικαστηρίου για τον ε, περιορισμό των ελευθεριών των ε, ε, γυναικών μουσουλμάνων. Δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση του δικαστηρίου. Θα ήθελα απλώς να πω ότι εμείς προσπαθούμε πάρα πολύ σκληρά να ενθαρρύνουμε τα κράτη-μέλη αλλά και τον επιχειρηματικό κόσμο να προσφέρουν καλές ευκαιρίες για γυναίκες μετανάστες προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν. Ε, ξέρω ότι η συζήτηση αφορά κυρίως μουσουλμάνες γυναίκες, αλλά εγώ θα ήθελα να αναφερθώ γενικότερα στις γυναίκες στη ε, μετανάστευση. Διαπιστώνουμε ένα ενδιαφέρον φαινόμενο. Αυτές οι γυναίκες ε, μετανάστες είναι καλύτερες, ε, καλύτερα εκπαιδευμένες, έχουν καλύτερη μόρφωση από άνδρες που φτάνουν στην Ευρώπη, αλλά είναι πολύ λιγότερες οι δυνατότητες που έχουν για να εκμεταλλευτούν τη μόρφωσή τους ώστε να βρουν μια θέση εργασίας. Ε, διαπιστώνουμε ότι τα κράτη-μέλη ασχολούνται με διαφορετικό τρόπο με το θέμα αυτό και ξέρω ότι προσπαθούν πολύ σκληρά ε, προκειμένου να υπάρχουν αποτελεσματικά σχέδια ένταξης ε, τα οποία υπάρχουν ήδη στα κράτη-μέλη και ε, κυρίως σε χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο ποσοστό νεοφυχτέντων, αλλά δεν ξέρω αν αυτό οδηγεί και σε πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Κάτι τελευταίο για το γεγονός ότι δεν υπήρχε αρκετή φιλοδοξία για την άδεια μητρότητας. Ναι, πριν ε, ολοκληρώσουμε τις εργασίες ε, για τη δέσμη μέτρων ε, για τη συμφιλίωση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, εξετάσαμε αν μπορούμε να συμπεριλάβουμε κάποια στοιχεία από τη δέσμη μέτρων για την άδεια μητρότητας, αλλά πιστέψτε με, θα το είχαν μπλοκάρει πάλι τα κράτη-μέλη. Πρέπει λοιπόν να είμαστε φιλόδοξοι μεν, αλλά πρέπει επίσης να είμαστε και ρεαλιστές. Όσον αφορά τα όσα ρώτησε ο κύριος Ουρτασούν για την ε, κλιματική δικαιοσύνη, όπως σας είπα, προσπάθησα να εξορθολογήσω το θέμα της ισότητας των φύλων ώστε να συμπεριληφθεί σε όλες τις ε, δραστηριότητες τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν ξέρω αν, να σας πω αν υπάρχει κάτι πιστικό για την ε, κλιματική δικαιοσύνη και τη στρατηγική για ε, τις κλιματικές αλλαγές, αλλά ε, προσπαθούμε να έχουμε στοιχεία για τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια, αναφέρθηκε και εδώ σήμερα, γιατί έχουμε πολύ συγκεκριμένη άποψη για το πώς θα πρέπει να προστατεύονται οι ευάλωτοι πολίτες βάσει της νέας δέσμης μέτρων για την ενέργεια. Ε, για τους ευάλωτες ε, πολίτες, ε, στους, ε, μάλλον με τον όρο ευάλωτες πολίτες, κυρίως αναφερόμαστε σε γυναίκες, διότι είναι πολύ μεγάλο τμήμα των ανθρώπων που ζουν σε συνθήκες ένδια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολύ λυπάμαι που το λέω αυτό και έχουμε πολύ συγκεκριμένη ορολογία και διατύπωση και ζητάμε από τα κράτη-μέλη να ορίσουν ποιο είναι το ποσοστό τη ενεργειακή ένδυα και ποιες είναι οι ομάδες των πιο ευάλωτων πολιτών στα κράτη-μέλη που θα πρέπει να την χάνουν ειδική προστασίας. Αυτό λοιπόν καλύπτεται από τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια. Όσον αφορά τις μη νομοθετικέ προτάσεις για τις συμφωνίες οικογενειακού και επαγγελματικού βίου και το πώ θα χρηματοδοτηθούν, αυτό το οποίο θα κάνουμε πιο συγκεκριμένα είναι ότι θα προτείνουμε στα κράτη-μέλη να επανασχεδιάσουν όπου μπορούν τις στρατηγικές τους, ώστε να υπάρχουν περισσότερα κονδύλια από το Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο για τις κοινωνικές υπηρεσίες. Διότι ε, θεωρώ ότι τα συστήματα χρηματοδότησης αυτά δεν θα πρέπει να είναι άκαμπτα. Ε, τα προγράμματα αυτά σχεδιάστηκαν κάποια στιγμή το 2012 για τη συγκεκριμένη προγραμματική περίοδο και νομίζω ότι πρέπει ε, από καιρού καιρών να τα επανεξετάζουμε, λαμβάνοντας υπόψη νέες προτεραιότητες, νέες ανάγκες και να έχουμε και το απαραίτητο σθένος να ε, κάνουμε νέο σχεδιασμό των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Αυτό λοιπόν συστήνουμε στα κράτη-μέλη θα κάνουν βεβαίως ό,τι μπορούν προκειμένου να υλοποιηθεί, διότι είναι διαφορετική η κατάσταση σε κάθε κράτος μέλος, αλλά θα συμβουλεύσουμε, ε, όχι ε, με οδηγίες, αλλά θα τους δώσουμε συμβουλές τι ακριβώς να κάνουν, διότι ε, τα πάντα πρέπει να βασίζονται σε μια πολύ καλή ανάλυση κόστους ωφελείας και θα συστήσουμε στα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν τον υπολογισμό αυτό προκειμένου να ορίσουν το κόστος, αλλά και τα κοινωνικά και μακροοικονομικά ωφέλη. τα οποία θα πρέπει να αρκούν ως λογική για να επενδύσουμε τα χρήματα ε, σε συγκεκριμένε υπηρεσίε. Συγγνώμη που τα είπα έτσι περίπλοκα, αλλά έπεσα και εγώ μόνη μου στην παγίδα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τις απαντήσεις σας. Έχουμε ερωτήσεις από δύο μέλη. Οπότε θα ήθελα να δώσω το λόγο στην κυρία Πετήρ, παρακαλώ. Σύντομα παρακαλώ, μόνο έχετε μόνο 10 λεπτά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. E, iziskuje od nas veće napore koje moramo e, uložiti. E, Όσον αφορά την παραβίαση των δικαιωμάτων των γυναικών, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα προκειμένου να υπάρχει αξιοπρεπή εργασία για όλου του εργαζομένου και να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και καλή ισορροπία μεταξύ επαγγελματικού και ε, οικογενειακού βίου. Οι έρευνε απέδειξαν ότι ε, κατάλληλος χρόνος ξεκούρασης στη διάρκεια της ημέρας εργασίας μπορεί να μειώσει τους ψυχογονικούς κινδύνους όπως για παράδειγμα το στρες ε, και την υπερκόπωση. Οι εμπειρογνώμονες ε, για την προστασία στο χώρο της, ε, υγείας στο χώρο της εργασίας δημοσίευσαν κάποιες ανησυχητικές στατιστικές οι οποίες καταδεικνύουν ότι η κύρια αιτία απουσίας από την εργασία είναι μυοσκελετικά προβλήματα και επίσης ψυχοκοινωνικές ασθένειες και άγχος. Ε, και επίσης διαπιστώθηκε ότι η πρώτη αιτία του άγχους ε, ε, είναι η μεγάλη ημέρα εργασίας, και βλέπουμε ότι οι εργοδότες δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά διότι θεωρούν τα αίτια ε, του άγχους και των παθολογικών αυτών καταστάσεων οφείλονται στην προσωπική του ζωή και όχι στην εργασιακή. Ε, οι άνθρωποι αυτοί δουλεύουν τουλάχιστον μία ημέρα την εβδομάδα πάνω από 10 ώρες. Θα ήθελα να ρωτήσω το εξή, κυρία Επίτροπε. Τι μέτρα σκοπεύετε να λάβετε ώστε να υπάρχει όντω ισορροπία μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, να υπάρχει ευημερία των εργαζομένων και να μπορούν να έχουν χρόνο εργασίας, ο οποίος θα είναι αξιοπρεπής και όπως επίσης και η μέρα ξεκούρασης όπως ε, ε, είναι συνήθως η Κυριακή. Για τον σχολιασμό των νομοθετικών και μη νομοθετικών μέτρων, πιστεύω ότι είναι αρκετά φιλόδοξα. Ήδη είπατε κυρία Επίτροπε πως δεν θα είναι εύκολο για κάθε μεμονωμένο κράτος μέλος να εφαρμόσει τα μέτρα αυτά. Φυσικά κάποια κράτη-μέλη έχουν ακόμα πιο φιλόδοξες προτάσεις. Αλλά πιστεύω πως αποκείται στα επιμέρους κράτη-μέλη να ασχοληθούν με το ζήτημα. Μου αρέσει η πρότασή σας όσον αφορά την γονική άδεια, την πατρική άδεια. Επίσης συμφωνώ με τις περιόδους μη μεταφοράς, μη μεταβίβασης, επειδή είναι σημαντικό για τα παιδιά και πρέπει να τονίσουμε το θέμα. Είναι πολύ πιθανό πως κάποια κράτη-μέλη θα αρνηθούν να ανταποκριθούν στο καθήκον αυτό, αλλά πιστεύω πως θα πρέπει να καταλάβουν πως πρόκειται για έναν τρόπο υποστήριξης των οικογενειών και των γονέων. Μου αρέσει η πρότασή σας για πενθήμερη άδεια σε περίπτωση που ένας συγγενής σας είναι άρρωστος Το ίδιο ισχύει επίσης για την άδεια ασθενείας, επειδή αυτό που μας λείπει στην κοινωνία μας είναι περισσότερα παιδιά και καλύτερη φροντίδα, όχι μόνο των παιδιών, αλλά επίσης των ηλικιωμένων μελών των οικογενειών μας. Μιλήσατε για 370 δισεκατομμύρια ευρώ κατά προσέγγιση που χάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν οι γυναίκες δεν εργάζονται. Αλλά δεν μιλούμε για τις απώλειες που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω του γεγονότο πως παιδιά δεν γεννιούνται. Και μέχρι η κοινωνία μας να σεβαστεί την εργασία που σχετίζεται με την φροντίδα των παιδιών, δεν θα έχουμε μόνο το μισολογικό χάσμα, αλλά επίσης ένα χάσμα παιδιών. Και αυτό πιστεύω πως τουλάχιστον για μένα είναι το πιο σοβαρό πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γνωρίζω πως η εργασία σας δεν είναι εύκολη, δεν θα είναι εύκολη για να προωθήσει όλα αυτά τα ζητήματα, αλλά κάτι που θα ήθελα να πω, στο οποίο αναφερθήκατε επίσης, επειδή υπάρχει μια κάποια ανισορροπία εδώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σέβεται τη φροντίδα παιδιών ως αξία η οποία θα πρέπει να γίνεται σεβαστή. Και αυτό ισχύει επίσης για την ιδιότητα του γονέα αλλά είδα ότι καλύψατε κάποια θέματα στην πρότασή σας. Επιτρόπος, ευχαριστώ πολύ για τα, και τις παρατηρήσεις σας σχετικά με το χρόνο εργασίας. Έχουμε τώρα τη δρομολόγηση των διαπραγματεύσεων των κοινωνικών εταίρων για την οδηγία για, τους, για τις ώρες εργασίας. Ανήκει στο θεματοφυλακείο Τάισεν. Επίσης έχουμε την οδηγία για τις ώρες εργασίας που είναι ανοιχτή για διαβούλευση, για συζητήσεις αλλά δεν είναι, είναι στην αρμοδιότητα του Μαριαν Τάισεν It Της Μαριάν Τάισεν, συγγνώμη, αρχίσαμε στις 26 Απριλίου σύμφωνα με τους κανόνες θα διαρκέσει 8 εβδομάδες ανοιχτή για διαβούλευση λοιπόν η οδηγία συμφωνώ μαζί σας πως είναι ακραία η επιβάρυνση και με αυτή τη δέσμη μέτρων για ευέλικτες σχέσεις εργασίας προσπαθούμε να προσαρμόσουμε το πλαίσιο στον 21ο αιώνα καθώς ήδη πολλές θέσεις εργασίας επιτρέπουν καλύτερες συνθήκες καθώς απαιτούνται προσπάθειες για ανθρώπους που προσπαθούν να συνδυάσουν την οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή και είναι σημαντικό για αυτούς να λαμβάνουν την προσφορά μια τέτοια δυνατότητα. Γι' αυτό και πιστεύω πως, είναι, πιστεύω πως μπορούμε να βελτιώσουμε εν μέρη την κατάσταση κάποιου μέρους της κοινωνίας μας με αυτή τη δεσμή μέτρων για τον συνδυασμό ιδιωτικής και επαγγελματική ζωής όσον αφορά την ερώτηση για το χάσμα παιδιών αν υπάρχει ναι φυσικά υπάρχει Ε, είναι ένας από τους λόγους για τον οποίο δρομολογήσαμε τη δέσμη μέτρων για τη γονική άδεια. Δεν πιστεύω πως αν οι άνθρωποι πληρώνονται ή όχι είναι τόσο σημαντικό τόσο σημαντικός αποφασιστικός παράγοντας για αυτούς στην επιλογή τους αν θα κάνουν παιδιά ή όχι. Αλλά μπορεί ίσως να είναι παράγοντας για κάποιους, για κάποιους άντρες να μοιραστούν τις ευθύνες με τις συζύγους τους και επίσης θα μπορούσε να αποτελέσει παράγοντα για γυναίκες οι οποίες πρέπει να κάνουν την φοβερή αυτή επιλογή του είτε να κάνουν μια επαγγελματική σταθειοδρομία είτε να κάνουν παιδί. Γι' αυτό και προσπαθούμε να ανοίξουμε χώρο για μια καλύτερη λήψη αποφάσεων και πιο ανώδυνη. Αυτή είναι η συνεισφορά μας επί του παρόντος. Ε, πιστεύω πως το Κοινοβούλιο σχετικά με, το, με τη δέσμη μέτρων αυτή θα περιμένω πιο θετικές αντιδράσεις από ό,τι από τα κράτη-μέλη, αλλά θα εργαστώ πολύ σκληρά για να έχω πιστικά επιχειρήματα, έτσι ώστε η δέσμη μέτρων αυτή να εγκριθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Πρόεδρος. Κυρία Επίτροπε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψή σας, για την παρουσίασή σας, για τις απαντήσεις σας και τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους όλων μας. Ευχαριστώ και εγώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ήταν το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συνεδρίαση. Θα τα πούμε αύριο στις 9 το πρωί. Θα αρχίσουμε με τη συνεδρίαση των συντονιστών και στις 9.30 με τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ πολύ.